Uh, uh, could I... Uh, Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, ώστε να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Good. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω θερμά στην απογευματινή συνεδρίαση. Έχει περάσει και κάποιος ε, καιρός από τότε που συναντηθήκαμε τελευταία φορά. Είχαμε και την Τυρκουάζ εβδομάδα. Όπως γνωρίζετε κάποιοι από εμά πήγαν σε μία επιτροπή στην Ινδία, μία Επιτροπή για να διαπιστώσουμε τι, τα καθέκαστα. Βλέπω η κυρία Ράπτη είναι εδώ. Ε, ήταν μια αποστολή που ήταν πολύ επιτυχημένη, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε και μια μικρή έκθεση της ε, ε συνεδρίασης με κάποια κόμματα και από τον τύπο από την συνέντευξη τύπου και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε και μια πλήρη συζήτηση με τα μέλη που πήγαν στο μέλλον. Ε, θα χαρούμε να ακούσουμε και τις απόψεις σας ούτως ή άλλως το να ταξιδέψει κάποιος ε, στην Ινδία στα πλαίσια της ευρύτερης προσέγγισης που κάνουμε για τις επιπτώσεις της εσωτερική αγοράς στην παγκόσμια οικονομία ήταν κάτι το οποίο ήταν ευπρόσδεικτο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές που το σκέφτηκαν και συμφώνησαν με αυτό. Ε, νομίζω ότι εκμεταλλευτήκαμε απόλυτα την ευκαιρία που μας δόθηκε. Επίσης, θα σας πω τις επόμενες εβδομάδες, ε, διότι όπως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς προσεκλήθην από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχω στη δεύτερη τριμερή σύνοδο για την ασφάλεια των εμπορικών προϊόντων που θα γίνει μεταξύ της Επιτροπής Ασφάλειας Προϊόντων ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της, ε, του Κινέζικου Ινστιτούτου Ποιοτικών Προδιαγραφών που συζητήσαμε, συναντήσαμε κάποιοι εξημών όταν πήγαμε στην Κίνα το 2008. Έγινε και μια συζήτηση πριν από δύο εβδομάδες. Σας έχει διανεμηθεί και μια δήλωση στο νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο πρόοδο. Είναι λίγο πιο ανοιχτή στην ανταλλαγή πληροφοριών η Κινέζοι εταίροι μα και στη διαδικασία αυτή. Και η κυρία Τάρεμπαουμ, που είναι η πρόεδρο από πλευρά των ΗΠΑ τη ε, αντίστοιχη επιτροπή, και αν θυμάστε καλά, ήρθε να μα μιλήσει το Μάιο, μου ζήτησε να διαβιβάσω τι ευχέ τη ε, και είναι χαρούμενοι που εξακολουθεί να συνεχίζεται αυτή η ενεργός συνεργασία με αυτούς. Νομίζω ότι και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για την Επιτροπή μας. Αυτά λοιπόν ως ενημέρωση για τα όσα κάναμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα να εγκρίνουμε την ε, ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα για όσους από εσά ε, θα ήθελαν να γνωρίζουν, η ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Βάιας ε, Γκέρμπερ αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε διότι το Συμβούλιο δεν είχε ακόμα χρόνο να συναντηθεί και να επιβεβαιώσει επισήμως την αποδοχή της πρότασης και κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να συζητηθεί και να ψηφιστεί το θέμα στην Επιτροπή μας πριν λάβουμε την επίσημη επιστολή από το Συμβούλιο η οποία θα επιβεβαιώνει ότι έχονται τις προτάσεις. Μόλις τη λάβουμε θα προχωρήσουμε το θέμα και θα το ψηφίσουμε. Έχουμε μια σημαντική συζήτηση με την κυρία Στάιλερ για την ε, εμπορία ε, των δομικών προϊόντων και το χρονοδιάγραμμα και από εκεί και πέρα μια ψηφοφορία που θα γίνει στις 3.30. Ε, σας έχουμε ζητήσει να φέρετε και τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε και Κατόπιν θα ξεκινήσουμε και τις εργασίες για την ε, ε, γνωμοδότηση του κυρίου Τιόν για ο Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκά Διπλώματα χνίας. Να σας πω τώρα και κάποιες ε, τεχνικές λεπτομέρειες. Καταρχάς η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και επίσης επειδή υπάρχει ε, γρήπη στη σουηδική κοινότητα και στους σουηδικούς διερμηνείς, δεν θα έχουμε σουηδική καμπίνα σήμερα. Μπορείτε να μιλήσετε, αλλά δεν μπορείτε να ακούσετε σουηδικά. Ε, δεν είναι κάποιο Σουηδό συνάδελφο εδώ, αλλά οποιοδήποτε περίμενε να ακούσει Σουηδικός, ε, Σουηδικά, δυστυχώ, δεν μπορούμε να έχουμε τις εξαιρετικές υπηρεσίες διερμηνίας, ε, όπως συνήθως λέει ο πρόεδρο. Όσοι οι υπόλοιπε καμπίνες λειτουργούν κανονικά. Να προχωρήσουμε τώρα στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Εξέταση τροπολογιών για τα δομικά προϊόντα και τη σχετική οδηγία. Ε, ξέρω ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην μετάφραση των τροπολογιών. Νομίζω ότι η συγγήτρια, ε, αλλά έχω λάβει και εγώ ένα σημείωμα για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, αλλά θα αφήσω την ίδια την συγγήτρια να σας πει για το θέμα αυτό. Να σας παρουσιάσω και την άποψή της για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και μετά έχουμε και τους κοιόδης εισηγητές ε, που θα μιλήσουν. Ο κύριος Μπουσόη δεν ε, είναι εδώ. Ο κύριος Σαλβίνη δεν είναι εδώ επίσης. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα ακούσουμε και τους κοιόδης ηγητές όσους είναι εδώ. Κύριε Στάιλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδης εισηγητές και θα ήθελα να σας πω ότι ε, λυπάμαι που δεν μπορείς να ε, συναντηθούμε ε, με τους, τους σκιώδεις από όταν υπάρχει η διερμηνή ή μετασφαλισμένη μετάφραση και γι' αυτό ε, εάν δεχτούν οι συντονιστές τώρα θα ήθελα να συναντηθούμε στις 22 του μηνός το βράδυ για να μπορέσουμε να συζητήσουμε επί της μεταφράσεως. Ε, ξέρω ότι το χρονοδιάγραμμα μας ήταν διαφορετικό, αλλά λόγω της φύσης ε, του εγχειρήματο και ε, του κειμένου που προσπαθούμε να καταρτήσουμε, έχουμε ως τις 22 του μηνός καιρό να δούμε πού συγκλίνουν οι απόψεις μας και πού πιστεύουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει σχετικά με τις τροπολογίες. Όσον αφορά τη συνάντηση της 22ης του μηνός ε, ε, εφόσον ε, έπρεπε να απαντήσουμε σε ορισμένα θέματα. Μπορέσαμε ήδη να βρούμε σημεία στα οποία συγκλίνουμε και υπάρχουν διάφορα προβλήματα επί των οποίων δεν έχουμε πρόβλημα. Βέβαια όσον αφορά τις συγκεκριμένες τροπολογίες πρέπει ακόμη να τις επεξεργαστούμε. Δεν θέλω να προκαταλάβω αλλά θα τις κοιτάξουμε την επόμενη εβδομάδα και προσπαθούμε να βρούμε ε, κοινά σημεία στα οποία συμφωνούμε και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν ε, να πω στους συναδέλφους ότι αν θέλουν να σχολιάσουν τα δικά του συγκεκριμένα θέματα επί των τροπολογιών βλέπω ότι η κυρία Ρούδ και ο κύριος Μάιρς είναι εδώ, εγώ είχα ήδη δύο φορές ε, την ευκαιρία να σχολιάσω τα δικά μου θέματα, οπότε θα ήθελα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να τους δώσω τώρα το λόγο για να σχολιάσουν αυτοί τα θέματα που ίσως θέλουν να θίξουν. Ευχαριστώ, κυρία Στάιλερ. Αντιλαμβάνομαι σε ποια κατάσταση βρίσκεστε και ελπίζω ότι με την ε, τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ε, θα μπορέσουμε ε, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, τη παρουσία τους. Και είμαστε πολύ, έχουμε πολύ κατανόηση για τη θέση σας. Ε, δέστε λοιπόν τι θα κάνετε με τους χειώδεις εισηγητές και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τον κύριο Μάε του ΕΛΚ. Μετά θα ήθελα και εγώ να κάνω ορισμένα σχόλια εκ μέρους της σκιώδης εισηγήτριάς μας της κυρίας Κλάρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μάιρς. Συμφωνώ με την ε, εισηγήτηρια η οποία είναι πολύ επιμελή στην επεξεργασία του θέματος αυτού. Δεν είναι όμως δυνατόν τόσες πολλές τροπολογίες και τόσο εκτενείς τροπολογίες να ε, τις επεξεργαστεί κανείς εάν δεν τις έχει στην γλώσσα του. Γι' αυτό και μεταθέσαμε τις ημερομηνίες. Παρόλα αυτά στην προηγούμενη κοινή συνεργασία με τους χιώδεις εισηγητές μπορέσαμε να προχωρήσουμε διάφορα θέματα όσον αφορά τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και προσεγγίσαμε τις θέσεις μας ακόμη και αν δεν έχει βρεθεί ε, ε, μια συμβιβαστική λύση. Είναι όμως ακόμη πολλά θέματα που εκκρεμούν και γι' αυτό στο μέλλον θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα θέματα αυτά. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση κύριε Πρόεδρε και το πιο βασικό είναι ότι και στην έκθεση αυτή επανέρχεται κανείς συνέχεια στο τι μέλη γενέστε περί του πρακτέου. Δηλαδή, ε, από το 1957 προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την κοινή αγορά, να την ανοίξουμε ε, και ε, θέλουμε ε, να υπάρχει απελευθέρωση της αγοράς. Άλλα θέματα έχουν προχωρήσει. Η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων και άλλα. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχή προσκόμματα τα οποία πρέπει να ε, ξεπεράσουμε και ε, γι' αυτό πολλές φορές οι αντιμετωπίσεις δεν είναι πολύ λογικές. Θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση διότι πιστεύω ότι όσον αφορά την ε, ψηφοφορία χαιρετίζω την έκθεση Ζουβά που ήταν εξαιρετική και με λίγες τροπολογίες όμως βλέπω ότι δεν θα απελευθερώσουμε τη διαφορά διαφήμιση αλλά θα την περιορίσουμε. Οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, ε, για κάθε τροπολογία στην ουσία. Να αναρωτηθούμε γιατί είμαστε εδώ. Δεν είμαστε για να περιορίζουμε, είμαστε για να απελευθερώσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο ε, κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν ονόματι του συναδέλφου Μπουσόη θα ήθελα να χαιρετήσω την επιμέλεια της ε, εισηγήτηριας και να την ευχαριστήσω ε, για τις προσπάθειές της. Έχουμε κάνει ε, ορισμένες συναντήσεις και προσεγγίσαμε τις θέσεις των πολιτικών ομάδων διότι η οδηγία την οποία επεξεργαζόμαστε είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για την βιομηχανία αλλά και για τον καταναλωτή με τους φιλελεύθερους υπάρχει μία συμφωνία για τη θέση που θα προβάλλουμε προς το Συμβούλιο ε, όσον αφορά την κατάσταση από τη σκοπιά την οικονομική και του καταναλωτή. Ε, γι' αυτό και στη συζήτηση με το Συμβούλιο είχαμε μία καλή βάση και ο κύριος Μπουσόη πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να κοιτάξουμε να καταλήξουμε σε μία σε έναν γερό συμβιβασμό διότι θα πρέπει να συνεργαστούμε κατά τρόπον ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή θέση στη δεύτερη ανάγνωση και να προωθήσει τις θέσεις του. Γι' αυτό και βάσει των συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα με τους σκιώδεις συζητητές, ο συνάδελφος Μπουσόη πιστεύει ότι είμαστε σε καλό σημείο για να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε η κυρία Ρούλε. Και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στάιλερ για την ε, καλή συνεργασία και όντως βοήθησε πολύ. Πρέπει όμως να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, με ενοχλεί στις τεχνικές συναντήσεις ότι ε, η, η, η τροπολογία συζητούνται μόνο σε επίπεδο εμπλεκομένων και όχι συνεργατών τους. Βλέπω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην τελευταία συνεδρία στι ορισμένε τροπολογίες και αυτό δεν είναι σωστό, διότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συζητήσει μαζί μας θα πρέπει να συνεννοηθεί με τους ευρωβουλευτές, να κλείσει ραντεβού με τους ευρωβουλευτές και όχι να τα συζητήσει με τους συνεργάτες τους διότι αυτή η οδηγία σχετικά με τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών είναι πολύ σημαντική και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε απλό επίπεδο συνεργατών διότι στο μέλλον δεν θα συμμετέχουν οι συνεργάτες μας σε θέματα πολιτικών, πολιτικού επίπεδου εάν αυτό είναι το αποτέλεσμα κάποια σχόλια από πλευρά μου, εξ ονόματο κυρία Μακλάρκ που κατέθεσε και τροπολογίε, αλλά να συνεχίσω και από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι τα θέματα που είναι πιο δύσκολα αφενός αφορούν πολύ μεγάλους οργανισμούς ε, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν μεγάλες παραγωγές σε μεγάλες εγκαταστάσεις αλλά ισχύουν και για πολύ μικρότερους ε, κατασκευαστές δομικών προϊόντων, ε, τα οποία ορισμένες φορές είναι φτιαγμένα ειδικά για ένα συγκεκριμένο κτίριο ή για κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία και που μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλους ε, τρόπους παραγωγής που, ή άλλα κομμάτια παραγωγής που μπορεί να έρχονται από πολύ μεγάλες βιομηχανίες. Πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο θα διευκολύνει τη λειτουργία της αγοράς, της ενίας αγοράς και σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε σαφή εφαρμογή υψηλών προδιαγραμμών, εναρμονισμένο στο βαθμό του δυνατού. Αλλά δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε περι, και μη ρεαλιστικά άχθη, κυρίω σε θέματα πληροφοριών προ του καταναλωτέ, σε περιπτώσει που δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία κατασκευή και νομίζω ότι κάποιες από τις προτάσεις να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές πληροφορίες που θα βασίζονται στο διαδίκτυο είναι ο καταλληλότερος τρόπος, διότι συνήθως αυτά είναι επαγγελματικά προϊόντα και ε, θα είναι πιο εύκολη πρόσβαση για όσους ενδιαφέρονται να ε, δουν ε, τα, τις πληροφορίες αυτές. Θέλουμε να έχουμε και κάποια σημεία επαφή. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνήσαμε στη γενικότερη δέσμη των μέτρων, το οποίο θα διευκολύνει και τη ζωή των μικρότερων επιχειρήσεων. Αυτά τα σημεία επαφή για τα προϊόντα θα βοηθήσει στα κράτη-μέλη να τα λειτουργούν αυτά σε συμφωνία ε, και με τα υπόλοιπα ε, προϊόντα ε, και τα σημεία επαφή για τα υπόλοιπα προϊόντα. Νομίζω ότι αυτά τα σημεία θα συζητήσουμε αργότερα. Και τέλος, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η οδηγία αυτή συνάδει πλήρως με όλα όσα έχουμε κάνει με τα πακέτα για τα προϊόντα ε, και για την εποπτεία της αγοράς και να υπάρχει πλήρη συσχέτιση, να μην δημιουργηθεί καμία σύγχυση. Αυτό νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία. Και όσον αφορά τώρα την εφαρμογή, και πάλι γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, κυρίως ως προς τη συσκευασία, έχουμε να κάνουμε ασυνεπή, με ασυνεπή εφαρμογή. Σε κάποιες χώρες μέλη δεν υπάρχουν οι πόροι για να εφαρμοστούν καταλήλως ε, οι διατάξεις και θα ήθελα να σας ζητήσω να μην δημιουργήσετε υπερβολικό άχθος για τις ε, αρχές εποπτείας της αγοράς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η οδηγία θα είναι αποτελεσματική. Νομίζω ότι το Συμβούλιο τα έχει λάβει υπόψη του αυτά τα σημεία. Υπάρχουν κάποιε πολύ σημαντικέ βελτιώσει στο έγγραφο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τι πρακτικέ πτυχέ ε, εφαρμογής αυτής της οδηγίας επιτόπου και στην οικοδομή, όχι στι συζητήσει μα εδώ στην Επιτροπή. Εκεί θα αποδειχθεί κατά πόσον είναι αποτελεσματική η οδηγία στι ε, διαφορετικέ ε, συνθήκες που επικρατούν σε σχέση με τα άλλα προϊόντα που συζητούμε. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Η κυρία Γκέπχαρτ είναι στον κατάλογό μου. Κυρία Γκέπχαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κατρίν για την πάρα πολύ καλή δουλειά την οποία ναι έκανε. Είναι μια πολύ τεχνική ε, έκθεση αλλά συγχρόνως πολύ πολιτική και δεν είναι εύκολο στον τομέα αυτό να βρει κανείς τις σωστές λύσεις διότι οι μεγάλες βιομηχανίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τελείως αντικρουόμενες απόψεις και χρειάζονται και διαφορετικές απαντήσεις. Οπότε το να βρεθεί το σωστό μέτρο να βρεθεί ε, η σωστή μέση οδός δεν είναι κάτι τόσο απλό. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κατρίν Στάιλερ κατάφερε να βρει αυτή τη μέση οδό και γι' αυτό πρέπει να τη στηρίξουμε θέλω να διευκρινίσω κάτι άλλο σχετικά με την ερώτηση του κυρίου Μάιερ. Βεβαίως η ελευθερία είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικοί περιορισμοί. Αλλά και η ασφάλεια είναι πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δεν πρέπει να παραβλέπουμε και επίσης ε, και αυτό προβλέπει περιορισμούς. Ως εκ τούτου θα πρέπει αυτά τα μέτρα ασφαλείας των προϊόντων να έχουν ληφθεί υπόψη. Δεν είναι πολύ αυτό, απλό να λέμε ότι θέλουμε περισσότερη ελευθερία και λιγότερο περιορισμούς πρέπει να σκεφτόμαστε την ασφάλεια των προϊόντων, των χρηστών, των ανθρώπων που χειρίζονται αυτά τα προϊόντα και όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και νομίζω ότι η Κατρίν βρήκε μία πολύ καλή λύση στο θέμα αυτό και την θεστηρίζω για να προχωρήσει τη δουλειά της. Η κυρία Βάις Γκέρπερ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ καλό με πόσο δομημένο τρόπο και κατόπιν των ακροάσεων με πόσο ο καλές βάσεις έχει καταρτιστεί η έκθεση αυτή, αλλά σαν απλή ε, ευρωβουλευτής και σαν απλό μέλος στην αρμόδια επιτροπή θέλω να παρέμβω και να στηρίξω την κυρία Ρούλε, διότι άκουσα ότι υπάρχουν αυτές οι τεχνικές συναντήσεις με το Συμβούλιο και εγώ σαν απλό μέλος της Επιτροπής θέλω να ρωτήσω, συνηθίζει να υπάρχουν τόσο έντενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο πριν την ψηφοφορία. Μήπως αυτό οδηγήσει, οδηγεί ότι θα απεμπολίσουμε ορισμένες θέσεις μας ε, πολύ νωρίς. Θα είναι λοιπόν πολύ βασικό να ε, υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις και ε, όσον αφορά τα θέματα στα οποία συμμετέχω στηρίζω αυτά που είπε η κυρία Ρούιλε. Επίσης θα ήθελα να σας πω χωρίς να επισέρχομαι σε λεπτομέρειες ότι έχω τρία ουσιαστικά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι επειδή δεν είχα την προηγούμενη φορά μία σωστή απάντηση θα ήθελα μία αξιολόγηση της εισηγήτριας διότι ε, θέλω να μου σχολιάσει τα τα προβλήματα και τα θέματα των πολύ μικρών ε, επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά την ε, συγγραφή των υποχρεώσεων, διότι είμαι εκπρόσωπος της πολιτικής μου ομάδος και πρέπει να σας πω ότι πρέπει πάντοτε οι πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των κανόνων και επίσης χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες και εφόσον πρόκειται για υποπροϊόντα ε, υπάρχουν ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες και παράγουν αυτά τα προϊόντα και τα χρησιμοποιούν. Οπότε θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή και γι' αυτό δεν θα πρέπει ούτε να εξαιρέσουμε ε, γενικώ τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ούτε να υπάρξει ιδιαίτερη μνήμα μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις ή στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δεν προσέξουμε να υπάρξουν τα αναγκαία εχέγγυα. Ε, δηλαδή Πρέπει ε, να έχουμε εξασφαλίσει και αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Και γι' αυτό θα με ενδιαφέρει να ξέρω πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της κυρίας Στάιλερ με το Συμβούλιο. Όσον αφορά το άρθρο 6 ε, ε, σχετικά με την τροπολογία 97 που έχω καταρτήσει, νομίζω ότι και εδώ, όπως είπε και η κυρία Ρούλε και ο κύριος Σβάμπ, θα πρέπει ε, να υπάρξει ένας χαρακτηρισμός όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών κατά τρόπον ώστε ε, ο κατασκευαστής ε, να μην υφίσταται της ανταγωνισμού αν πρέπει να ψάχνει τα χαρακτηριστικά για κάθε στοιχείο. Επίσης όσον αφορά τα, τις επικίνδυνες ουσίες, τους οδηγίες για τις χημικές ουσίες. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Χάρμπορ, ε, δεν πρέπει να υπάρξουν επικαλύψεις εις ε, την ε, νομοθεσία και θα πρέπει να ισχύσουν τα ίδια που ισχύουν και στην άλλη οδηγία διότι ό,τι έχει προβλεφθεί στην ε, ε, οδηγία του Ριτς θα πρέπει και εδώ ε, να ισχύσει διότι διαφορετικά θα υπάρξουν επικαλύψεις. Σας ευχαριστώ εκ προημίου για την απάντηση που θα μου δώσετε. Δεν βλέπω κάποιο άλλο να θέλει το λόγο. Θέλετε... Ο κύριος Μάιερ. Äh, Πολύ σύντομα. Μιλήσαμε ε, επανειλημμένως για μία οδηγία. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος θα ρυθμίσει πολλά πράγματα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης λέγεται ότι τα εργοτάξια θα πρέπει να μην θέτουν σε κίνδυνο την, ε, ε, την ασφάλεια των ανθρώπων. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο και αυτό θα πρέπει να καλύψει καλύπτεται και από τα προϊόντα. Είναι σαφέστατο. Τώρα, αν αυτό βέβαια είναι, ε, συνάδεια απολύτως με ε, την ε, ασφάλεια των ατόμων είναι κάτι όπου θα με βρείτε πολύ επιφυλακτικό διότι εάν ας πούμε πρόκειται για ένα θέμα αν θα φοράει κάποιος εργάτης γάντια ή κάτι άλλο είναι διαφορετικό εδώ μιλάμε για εμπορία και όταν μιλάμε για εμπορία ποιονών προϊόντων διότι ε, και για το διαδίκτυο εγώ συμφωνώ κύριε Πρόεδρε αλλά καταρχώς θα πρέπει να έχουν διερευνηθεί τα προϊόντα προτού ξεκινήσει η κατασκευή και δεύτερον ε, υπάρχει ένα προϊόν το οποίο παραδίδεται ή στο εργοτάξιο όπου υπάρχουν νέα διαφορετικά και ο εργάτης πρέπει να βρει το σωστό προϊόν άρα εκεί χρειάζεστε, χρειάζεται σωστή σήμανση και άρα γι' αυτό θα πρέπει όλα να έχουν προβρεθεί τη στιγμή που φτάνει το προϊόν στο εργοτάξιο. Και τέλος μία διευκρίνηση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει συζήτηση περαιτέρω αν, ε, ε, ε, αν εδώ θα ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, αν ε, ε, ε, θέλουμε ένα άθραυστο γυαλί, δεν μας ενδιαφέρουν άλλα χαρακτηριστικά, μας ενδιαφέρει να είναι άθραυστο όπως πρεσβεύεται. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε τέτοιου είδους παρατηρήσεις και τροπολογίες. πρόεδρος. Και τώρα... Να ακούσουμε την άποψη του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Κατόπιν εσείς θα δευτερολογήσετε και να συνοψίσετε για να ολοκληρώσουμε. Ο κύριο Ζακ Φερτράσεν είναι εκπρόσωπο του Συμβουλίου και ο κύριο Αγίλες εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με των επιχειρήσεων. Το Συμβούλιο, πρώτα κύριε Φερτράσεν, θα ήθελατε πρώτα να μας πείτε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι και εγώ πρέπει να σταθώ στην ποιότητα αυτής της έκθεσης, της έκθεσης της κυρίας Στήλερ. Πρόκειται για έναν κανονισμό ο οποίος εκ πρώτη όψεω μπορεί να φαίνεται θέμα τεχνικό, τεχνοκρατικό, όμως όσο περισσότερο το μελετά κανείς, διαπιστώνει δεν έχουν έρθει τα πράγματα, είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό τεχνοκρατικό έγγραφο, έχει στοιχεία ε, οικονομικά αλλά και πολιτικά και γι' αυτό σε αυτό το έγγραφο καλύπτουμε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως το είπατε και το είπαν και άλλοι. Έχουμε κάποια δράση για τις ε, ΜΜΕ, για τις μεγάλες επιχειρήσεις επίσης και είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα επομένως ανάλογα με το μέγεθο της επιχείρησης. Υπάρχει και θέμα ασφάλειας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όμως το θέμα της καθαρής ασφάλειας, όπως και η οργάνωσή της στο επίπεδο της εργασίας, είναι θέματα τα οποία α, ρυθμίζονται αλλού. Και Πρόκειται για, φυσικά για θέματα επικουρικότητας. Και όπως επισημάνατε έχουμε τις μικροεπιχειρήσεις. Όπως ε, είπαν οι προγραλήσαντες. οπότε και τονίζεται το πόσο σημαντικέ είναι για τον ε, τομέα αυτή τη δραστηριότητα και επομένω είναι δυνατόν να ε, υπάρξουν και συμπληρωματικά μέτρα, όπω να υπάρχει ενημέρωση για όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα πρέπει επίση να ληφθεί υπόψη και για αυτή την διάσταση, ούτω ώστε κάποια επιχείρηση που εξάγει σε όλη την Ευρώπη θα θέλει αυτής εξ αρχής να έχει όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά μια μικρή επιχείρηση, μια επιχείρηση που κινείται σε τοπική αγορά, θα πρέπει να δούμε το κατά πόσον ενδιαφέρεται ούτω ώστε να δει όλους, όλους αυτούς τους κανόνες και, και πρότυπα γιατί ακριβώς ανάλογα με το μέγεθος εξαρτάται ότι ζητάει η επιχείρηση. Άρα όσον αφορά τις ε, κατασκευές υπάρχουν πάρα πολλοί κατασκευαστές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία τη μικρή επιχείρηση ή τη μικροεπιχείρηση. Και όλα αυτά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε τώρα διάφορες τροπολογίε. Ορισμένε εκ των οποίων θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ε, αφορούν γενικότερα θέματα, θέματα περισσότερο των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι τις μικρομεσαίες και μικροεπιχειρήσεις. Τε και τέλος, για όλες αυτές τις ε, που έχουν υποβληθεί, πρέπει να σας πω ότι είναι εντυπωσιακό το πόσες έχουν ε, υποβληθεί, το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρεται η Επιτροπή σας για αυτόν τον κλάδο των δομικών κατασκευών και για την προστασία του κατασκευαστού αλλά και του καταναλωτού. Όμως θα αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για να τις διεξέλθουμε όλες αυτές γιατί έχουμε από τις 22 του μηνός μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και δεν θα κάνουμε και πολλές συναντήσεις. 17 και 18 είχε κάτι προγραμματιστεί, το, το για τις 22 περίπου, άλλη μία συνάντηση και επομένως. Διαπιστώνω τώρα ότι θα γίνουν αυτές όλες οι συνεδριάσεις χωρίς να έχουμε τις τελικές εκδοχές αυτών των τροπολογιών. Επομένως, δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα έτσι επέβαλαν, αλλά όσο πιο πολλές συμβαστικές πρωτολογίες βρείτε, και έτσι κατέβει ο αριθμός των τροπολογιών, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε και εμείς να ασχοληθούμε καλύτερα, γιατί αν έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες, τότε υποχρεούμεθα να δουλέψουμε πολύ περισσότερο γρήγορα, για να μην μπω τίποτα χειρότερο στο γόνατο. Επομένως, και εσείς πλευρά σας καθώς είναι δυνατό, προσπαθήστε να τις ενοποιήσετε όσο γίνεται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επαφές διαπραγματεύσεις ανάλογα με την εντολή μας Harbor. Θα σε ευχαριστούμε για τη θετική σας αντιμετώπιση. Και μας εξηγήσατε και όλα τα θέματα τα οποία καίνε το Συμβούλιο ο κ. Σαγούλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Tout d'abord, euh, essayer de d'être sûr de ce que j'ai entendu. Η Ρούλ, μίλαγε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη δική σας Επιτροπή. Γιατί ε, διατύπωσε κάποιες επικρίσεις και εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για τη δική μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρούλ, ναι, μίλησα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο συζητείτε τις τροπολογίες και ήδη προσπαθείτε να βρείτε κάποιες λύσεις. Από τεχνικής πλευράς δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για τροπολογίες από πλευρά σας, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τους βουλευτές. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσω στα γαλλικά. Για να είμαι ειλικρινή μαζί σα, δεν καταλαβαίνω ακριβώ τι εννοείται, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την προβλόμου διαδικασία, έχει καταρτήσει ένα σωρό κείμενα και το τελευταίο αφορά κάποιε παρατηρήσει επί των θέσεων του Συμβουλίου. Ξεκίνησε με την ε, τροποποιηθήσα θέση επί τη βάση των θέσεων του Κοινοβουλίου. Η επίσημη μας θέση. Και στη συνέχεια προχωρήσουν διατύπωση τη θέση μα ε, όσον αφορά το καθένα από τα κείμενα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Πέραν αυτού, εμεί ανέκαθεν ναι, είχαμε την ίδια τοποθέτηση. Και το επανέλαβα πολλές φορές σε σχέση με τις τροπολογίες που τώρα συζητούμε. Είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι και ανοιχτοί γιατί έχουν προσπαθήσει να συμβάλλουμε με τρόπο επικοδομητικό και θετικό. Δηλαδή, πέραν των όσων επίσημα έχουν διατυπωθεί και εγγράφος και αυτών που απαιτεί η διαδικασία, για τις υπόλοιπες τροπολογίες είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Εκτός από ορισμένα θέματα τεχνικά επί του σημείου αυτού συμφωνώ μαζί σας. Βεβαίω και η πρόταση αυτή, όπως και κάθε ε, νομοθέτημα έχει στοιχεία πολιτικά, αλλά βέβαια και έχει και κάποια άλλα τεχνικά τα οποία είναι πάρα πολύ δυσνόητα. Οπότε και εμείς είμαστε στη διάθεση όποιου θέλει εξηγήσει και θα τις παράσχουμε. Μιλάμε για 183 τροπολογίες από ό,τι ξέρω και ήδη έχουμε τονίσει ότι υπάρχουν ένα σωρό τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν τον αφηγούν. Γιατί υπάρχουν εδώ αντιφάσεις εσωτερικές μεταξύ των επιμέρους τροπολογιών. Προσπαθώ να σας το ξεκαθαρίσω. Για, για, για καλό σας το λέω. Προσπαθώ επομένως να καταλάβω καλύτερα το ότι πιστεύετε τόσο ώστε να πάνε ακόμα τα πράγματα κατά την υπόλοιπη διαδικασία. Και άκουσα αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Μάιερ όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής Βεβαίω και για μια πρόταση που αφορά την εσωτερική αγορά. Βεβαίω Υπάρχουν και θέματα ασφαλείας, τα οποία σχετίζονται με το θέμα μας. Και αυτό ήδη προελέχθη και δεν αφορά τόσο τις ε, κατασκευές, το, το προϊόν, αλλά την εκτέλεση κάποιου έργου. Και αυτά τονίστηκαν και στο επεξηγηματικό υπόμνημα, το explanatory memorandum, Και όσον αφορά τα προϊόντα, υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαχειριστεί κανεί την υπόθεση, υπάρχουν πολλοί τρόποι ακόμα πιο αποτελεσματικοί, πέραν δηλαδή αυτού του κανονισμού, διότι είπαμε ότι κυρίω αφορά την εσωτερική αγορά και αυτή είναι η δική μα γραμμή πλεύση. Σα επαναλαμβάνω, κυρία Ρούλ, εάν θέλετε για δύο λεπτά και να τα πούμε εκτό αιθούση, ούτω ώστε να καταλάβω καλύτερα τη θέση σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Well, I don't want to, uh, I don't want to uh, have a procedural discussion on this particular... Δεν θέλω να ξεκινήσουμε συζήτηση επί της διαδικασίας για τη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί νομίζω το θέμα που έθιξε η κυρία Ρούλε αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι συγητές διαχειρίζονται τα τεχνικά τους θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί καλύτερα να μας πει αν συμφωνεί ή διαφωνεί με μια τροπολογία, αλλά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίζουν. Και όπως ε, κατέστησα φες, ε, παρά το γεγονό ότι είναι πολύ τεχνικό αυτό ο κανονισμό, ε, υπάρχουν πολλοί πολιτικά θέματα που το διέπουν και η διαχωριστική γραμμή είναι πολύ δύσκολη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που θέλησε να προχωρήσει το θέμα αυτό, διότι από τη δική μου την πείρα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να έχουμε όλους τους ευρωβουλευτές μαζί την κατάλληλη στιγμή και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ε, πολύ καλά τεχνικά θέματα, αλλά πάντα τα μέλη θα έχουν την άποψή τους. Κυρία Ρούλε, αν θέλετε να θέσετε αυτό το θέμα επί της διαδικασίας, θα το κάνουμε στη συνεδρία των συντονιστών, όπου με χαρά θα το συζητήσω, ε, αν θέλετε να καθορίσουμε ε, κάποια σαφέστερα πράγματα. αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορούμε να εξετάσουμε και πώς ε, λειτουργήσε και θα μπορέσουμε να μάθουμε και κάποια πράγματα για το μέλλον. Να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και λίγο το θέμα του χρονοδιαγράμματος, κυρία Στάιλερ, διότι βάσει των δικών μου πληροφοριών εσείς προτείνατε να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Σήμερα δεν θα ψηφίσουμε σαφώς. Η Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Οι συντονιστέ δεν το έχουν αποφασίσει. Ε, μπορείτε κάλλιστα να ε, το παρουσιάσετε, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σήμερα. Στι 22 Νοεμβρίου θα αποφασιστεί και θα πρέπει να δούμε και αν υπάρχει αίθουσα για να το οργανώσουμε. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να ε, ψηφίσουμε και την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή που νομίζω ότι είναι η τελευταία ε, ομάδα, εβδομάδα Επιτροπών πριν κλείσουμε για τα Χριστούγεννα. Να σας δώσω το λόγο λοιπόν για να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και να μας πείτε και τι θέλετε να γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε και τη δυνατότητα να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές ή δυνατόν να ψηφίσουμε στις 22 Νοεμβρίου, διότι νομίζω ότι έτσι... δεν ξέρω αν θέλω να το σχολιάσει και το Συμβούλιο, ε, αν ε, γίνει αργότερα από τις 22 Νοεμβρίου ψηφοφορείο, σημαίνει ότι θα είναι πιο δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον ε, επί Βελγικής Προεδρίας και πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι μπορεί να μην προλαβαίνουν στις 22, το καταλαβαίνω αλλά εγώ θα προτιμούσα να ψηφίσουμε στις 22 Οι συνάδελφοι περιέγραψαν πολύ καλά τις δυσκολίες, ε, το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τομέα που είναι πολύ διαφορετικός και έχει και μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση για όσα κάναμε σήμερα, όπως ε, και τη σημερινή συνεδρίαση που δεν θα ψηφίσουμε, ε, θα παρακολύσει τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να ψηφίσουμε στις 22. Κάποιοι συνάδελφοι έθεσαν ερωτήσεις για την έκθεση να ε, υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι το θέμα για τις επικίνδυνες ουσίες ήταν απλώς θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση και απλώς την ξαναπαρουσιάσαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε από το πουθενά, είναι η αρχική μας θέση ως Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και τις σχετικές τροπολογίες. Νομίζω ότι η κυρία Βάισμπεργκερ ανέφερε τα θέματα αυτά στη συνεδρίαση στις 22 Οκτωβρίου. Προσπαθούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό δεν έχουμε ακόμα καθορίσει καλά τι συμβαστικέ μα προτάσει. Ε, θα μπορούσα κάλλιστα να σα πω τι σκοπεύουμε να κάνουμε και στην αυριανή συνεδρίαση με τους κοιόδης ηγητές θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε πού υπάρχει συμφωνία, πού υπάρχει διαφωνία και πού είναι σαφεί οι διαφορέ μα και α ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στι 22 Νοεμβρίου. Τέλο, γνωρίζω ότι ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μικροεπιχειρήσεις και αυτό είναι στο άρθρο 27 αυτό έχει να κάνει και με τη διαφορά μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Στις μικροεπιχειρήσεις νομίζω ότι έχουμε την ίδια άποψη με τον κύριο Μάγερ. Μιλάμε για κάτι μικρό που κάνει κάτι ε, πολύ συγκεκριμένο, ενώ υπάρχουν άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν ε, πολύ μεγάλη παραγωγή, πολύ τεχνική και είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα θέματα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε και νομίζω ότι είμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση και οι αυριανή συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική. Να καθησυχάσω δέτε και την κυρία Ρούλερ, η τεχνική συνεδρίαση δεν ε, είχε καμία πολιτική συζήτηση, ήταν ε, απλώ μια συζήτηση για τεχνικά θέματα, δεν αποφασίσαμε τίποτα πολιτικό. Αύριο στη συνεδρία, τη συγγήτρια με του κοιόδη συγγητές θα είναι η πιο σημαντική συνεδρίαση που θα κάνουμε, διότι θα συζητήσουμε και του συμβιβασμού που θα παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ τους και όδες Περιμένω να ψηφίσουμε στις 22 ε, στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Thank you I think as far as the, um, Ευχαριστώ κύριε Στάιλερ. Για τις 22 Νοεμβρίου νομίζω ότι πρέπει να πάρω και επισήμως έγκριση από τους συντονιστές. Ε, θα σας αποστείλουμε και σχετικό σημείωμα. Ελέξαμε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μια αίθουσα στις 22 Νοεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα για να ψηφίσουμε. Δεν βλέπω κάποιον να έχει αντιρρήσεις από τους συντονιστές, οπότε μάλλον αυτό θα κάνουμε, αλλά πρέπει να περάσουμε από την τυπική διαδικασία επιβεβαίωσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς και τους κοιόδης ηγητές και την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας διαβεβαιώσω δε ότι δεν θέλουμε να καθοστερήσουμε καθόλου το θέμα αυτό, απλώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον θέλουμε να εξετάσουμε διεξοδικά όλες τις τροπολογίες. Να ευχαριστήσω και την κυρία Στάιλερ για την ε, πάρα πολύ σημαντική και εντατική δουλειά που κάνει. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία, μόνο μία για σήμερα. Η κυρία Βάισμπεργκερ είναι εδώ. Εν τη απουσία σας κυρία Βάισκέρπερ, εξήγησα γιατί δεν είναι το θέμα σας στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Briefly. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Ε, ήδη ελέγχθη ότι το Συμβούλιο δεν έχει συμφωνήσει ακόμη και περιμένουμε. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές οι οποίοι στήριξαν ε, τις ε, προτάσεις του Κοινοβουλίου και τις συμβιβαστικές ε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να απαλείψουμε ακόμη περισσότερο τη γραφειοκρατία και θα συζητήσουμε στο τέλος του μηνός στην Επιτροπή για να ψηφίσουμε και το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εργασία σας επ' αυτού. Ας προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία και θα ήθελα όσοι έχουν τις ε, κάρτες τους ψηφοφοριών να με βοηθήσουν να κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε εάν ε, έχουμε απαρτία. Ε, ζητώ καταρχήν από το ΕΛΚ να ψηφίσουν όλοι όσοι είναι μέλη του ΕΛΚ. Έχουμε 31 άτομα, εκ των οποίων 11 θα ψηφίσουν. νομίζω ότι 13 είναι όλοι. Όχι, εντάξει. 13. Τώρα παρακαλώ τους σοσιαλιστές να ψηφίσουν όπως θέλετε. Μέχρι στιγμής ε, είναι 6. Έχετε τις κάρτες σας ψηφοφορίας. Βλέπω 10. Ε, ε, βλέπω, Εύελιν, ότι έχετε 10. Τώρα είμαστε 9. Δεν δουλεύει η κάρτα. Άλλαξε θέση. Ε, θέλουμε να μπορεί να βοηθήσει η Προεδρία. Λοιπόν, ε, νομίζουμε ότι είσαστε 10. Βλέπω τέσσερις ε, φιλελεύθερους, τρεις πράσινους, είμαι και εγώ εδώ και υπάρχει και ένας ανεξάρτητος. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε ε, θα ήθελα να χαιρετήσω τους ε, επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν την ώρα της ψηφοφορίας και θέλω, ελπίζω να περάσετε καλά την ώρα των ψηφοφοριών μας. Λοιπόν, κύριε Ζουβάν, θέλατε κάτι να πείτε προτού προχωρήσουμε στην ψηφοφορία της εκθέσεώς σας. Ναι κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε πάρα πολύ σύντομα. Μέσω της εκθέσεως αυτής ήθελα να βρω μία σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να έχουμε ισχυρή ε, διαφημιστική βιομηχανία στην Ευρώπη για να μπορέσει να στηρίξει την ε, αγορά ε, και να προασπίζει τα δικαιώματα όματα του καταναλωτή. Ε, έχουμε προχωρήσει καλά, έχουμε πολλές συμβιβαστικέ λύσεις, το θέμα είναι σημαντικό και πολλές φορές θα δούμε πού υπάρχουν διαφορές ε, διότι οι διαφορές ε, είναι μεταξύ πολιτικών ομάδων και έτσι αυτό δείχνει πόσο πολύπλοκο και πλούσιο είναι το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ζουβάν. Νομίζω ότι απλώς πρέπει να ελέγξουμε και πάλι τον αριθμό των σοσιαλιστών για να δούμε ότι λειτουργούν όλες οι θέσεις σας. Για να δούμε, θέλετε να ψηφίσετε όλοι οι σοσιαλιστές τώρα παρακαλώ. Ωραία. Έχουμε 10 τώρα. Λίγη ψηφοφορία. Οπότε, μπορεί να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα μηχανήματα μέχρι το τέλος. Ε, εδώ είναι η πρώτη συμβαστική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα προχωράμε στην τροπολογία 34 της κυρίας Τούρεν. 37. Ε, Ε, η διαγραφή του κυρίου Ροσφόρ υπέρ κατά 38 του κυρίου Ζουβά υπέρ κατά εγκρίνεται του κυρίου Πουπάκη η τροπολογία αποσύρεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα βρισκόμαστε στην 43 του κυρίου Ζουβά, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 του κυρίου Μπουζουτήλ, υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 υπέρ και 11 κατά. Τώρα προχωρώ εις ε, την τροπολογία 45 της κυρίας Ιβάνοβα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 47 της κυρίας Ιβάνοβα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και η τροπολογία 48 του κυρίου Ζουβάν σαν προσθήκη, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49 της κυρίας Ιβάνοβα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50 του κυρίου Ζουβάν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην 55 του κυρίου Διόν υπέρ αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 55. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, λίγη. Εγκρίνεται 18 υπέρ, 15 κατά. Προχωράμε στη συμβιβαστική 4 του κυρίου Ζουβέν και άλλων υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 59 του κυρίου Ζουβέν και Παντσέρη. Υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τροπολογία 59. Ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίθηκε 24 ε, υπέρ, 8 κακά και μία αποχή. Τροπολογία 60. Μέγερ ε, Σβάμπ Σόμερ υπέρ ηλεκτρονικά νομίζω. Ξεκινά. Με συγχωρείτε, εφόσον εγκρίθηκε η 59, προχωράμε στην 14 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και μετά έχουμε ένα δεύτερο τμήμα της τροπολογίας ε, της Επιτροπής Γυναικών που βλέπετε εδώ, δεύτερο μέρος, ε, χωριστή ψηφοφορία, ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά, ξεκινά. Παραγράφος 8β, νέων, ε, τροπολογία γυναικών, ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. απερίφθη 15 υπέρ 18 κατά. Τροπολογία της Επιτροπής Γυναικών Υπαριθμό 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και προχωράμε τώρα στην 66 του κυρίου Ροσφόρ. Ηλεκτρονικά. Η τροπολογία 66 του κυρίου Ροσφόρ. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίθηκε 16 υπέρ, 15 κατά και 2 εποχές. Προχωράμε στην συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 70 των κυρίων Λάιον και κυρίας Παρβανόβα. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 70 ξεκινά. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά θέλω να είμαι βέβαιος. Λίγη. Βεβαίως, 25 ε, κατά και 8 μόνο υπέρ. Συμβιβασική 7 ε, ε, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 Τον ε, Λιέμ Χόγνο και Παντσέρι. Ε, ηλεκτρονικά. 73 ξεκινά. Λίγη. Απερίφθη 14 υπέρ, 17 κατά και 2 αποχές. 74 της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ κατά απερίφθη 75 ε, και 76 ταυτόσημες ε, ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 77 της κυρίας Ιβάνοβα υπέρ κατά εγκρίνεται 78 του κυρίου Διόν προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Αλλά στο ελέγξουμε. Ήταν κάπως ασαφές. Μιλάμε για την τροπολογία 78 σαν προσθήκη. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη εγκρίθηκε 21 υπέρ και 12 κατά. Παράγραφος 15. Τροπολογία 79 Μακλάρκινγκ. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 80 του κυρίου Μότι. Εφόσον απερίφθη 79 υπέρ. Ε, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε για την τροπολογία 80 του κυρίου Μότι. Λίγη. Ερίφθη με 15 ε, υπέρ και 18 κατά. Η κυρία Τούρνεν, ε, τροπολογία 81, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 82 της κυρίας Ιβάνοβα. Υπέρ. Ηλεκτρονικά νομίζω καλύτερα. Μιλάμε για την ε, τροπολογία 82, ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Ε, ε, υπερψηφίστηκε 21 υπέρ 10 κατά. Ε, συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τώρα πάμε εις συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην 92. Μίστερ Τσέγκ Παγκάρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 Μότι ως προσθήκη. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 94 Ζουβά Όχι, καλύπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπία 14. Υπέρ. Συμβαστική τροπολογία 14. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρα περνάμε στα θέματα τα οποία καλύπτει ο συμβασμός. Καταρχάς, τροπολογίες 96, 97, 98 που είναι διαγραφή. 96, 97, 98 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 99, 100, 101, 102, 103 και 104 καταπίπτουν, επομένως πάμε στην 105. 105 από την κυρία Έσια. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 107 και 108 που είναι πανομοιότυπες, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Όλες οι υπόλοιπες καλύπτονται από τη συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία 15, παράγραφος 17, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 115 του κυρίου Μότι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116. Κατά τμήματα. Κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ και έχετε το σημείο που χωρίζεται. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 14 υπέρ 19 κατά. Συμβαστική τροπή απολογία 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 118 από του κύριο Πουπάκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. 119 του κυρία Τάιλερ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σαφώς. 120 του κυρίου Μότη. Καταπίπτει, συγγνώμη. Πάμε στην 123. 123 Ρόσφορ. Συγγνώμη. ΦΕΜ 4. Δεύτερο και τρίτο τμήμα της τροπολογίας. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά τους εδώ. Δεύτερο και τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 123 του κυρίου Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 124 μότι. Υπέρ. Νομίζω ότι θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 124 του κ. Μότη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. 125. Γκοκ Πατσέρι. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 126 της κυρίας Παπαδοπούλου. Άρχεται η ψηφοφορία για την 126 της κυρίας Παπαδοπούλου. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 130 λοιπόν. Λάιον Ροσφόρ Παρβανόβα, η κυρία υπέρ. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 130. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφι, 21 ψήφι υπέρ 11 κατά. 131 καταπίπτει. 132 από τις κυρίες Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επιτροπή Γυναικών 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επιτροπή Γυναικών 10 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Επιτροπή Γυναικών 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επιτροπή Γυναικών 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γυναικών 1. Το πρώτο τμήμα. Μόνο η φράση που έχετε εδώ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Επιτροπή Γυναικών 2. Υπέρ. η ηλεκτρονική επαλήθευση για την ε, τροπολογία αυτή. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 12 υπέρ 19 κατά. Επιτροπή Γυναικών 4, πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 13 υπέρ 19 κατά. Επιτροπή Γυναικών 5 υπέρ. Και πάλι μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Επιτροπή Γυναικών 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 12 υπέρ 19 κατά. Επιτροπή Γυναικών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. vote κατά πέρας ψηφοφορία, συγγνώμη, εγκρίνεται 18 υπέρ, 14 κατά. Επιτροπή Γυναικών 7. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται 14 υπέρ, 19 κατά. Επιτροπή Γυναικών 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψίφικατα. Πιτροπή κυνηγών 13. Άρχετε ψυχοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ 21 ψήφι κατά. Η Επιτροπή Γυναικών 13. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψυχοφοριας ψηφοφορίας. Μόνο 2 είναι υπέρ, 10 αποχές και 21 ψήφι κατά. Περνάμε λοιπόν στη συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ και πάλι θα κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 18. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Να περάσουμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 6. Για την αιτιολογική σκέψη α1 και πάλι ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 6. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, 2 αποχές. Τροπολογία 7. Διαγραφή. Υπέρ. Και πάλι θα κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 10 ψήφοι υπέρ, 23 κατά. Να περάσουμε τώρα στην τροπολογία 8 της κυρίας Μακλάρκιν, η οποία είναι κατά τμήματα κατόπιν ετήσεως του ΕΛΚ. Για το πρώτο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19 αιτιολογική σκέψη C υπέρ κατά, αποχές εκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 11. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Τροπολογία 12, Ηλιάνα Ιβάνοβα. Κύριε Ιβάνο, θα ήθελα να την αποσύρω, διότι είναι επανομοιότυπη με την επόμενη. Την αποσύρω λοιπόν. Η τροπολογία 12 αποσύρεται, λέει ο πρόεδρο. Θέλει κάποιο να καταθέσει ε, ε, ένσταση. Όχι. Η τροπολογία 13, η οποία είναι προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14, κύριο Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 στην αιτιολογική σκέψη τι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 20, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 25 που είναι από τον κύριο Ντεγιόν κατά τμήματα ψηφοφορία κατόπιν του ΕΛΚ. Ψηφίζουμε πρώτα το τμήμα 1 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Τμήμα 2 της τροπολογίας 25 υπέ, η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 26. Και πάλι κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 ψήφι υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 27 της κυρίας Παπαδοπούλου. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 27. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 ψήφι υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 28 και πάλι της κυρίας Παπαδοπούλου, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάλι. 18 ψηφί υπέρ, 15 κατά. On the final opinion, which I propose to take by electronic vote. Να ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικό στο κείμενο ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 30 ψήφοι υπέρ, μία κατά και δύο εποχές. Ευχαριστούμε κύριε Ζουβά. Σα ευχαριστούμε για τη δουλειά σας. And thank you very much, colleagues, for support. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την ψηφοφορία. Θα κάνουμε τώρα ένα διαλυματάκι, ένα-δύο λεπτά, να φύγει ποιος να φύγει και κατόπιν θα λάβει το λόγο ο κ. Δεγιόν. Αλλά παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως, ούτως ώστε να μπορούσαμε να συνεχίσουμε. παρακαλώ συνεχίστε την συζήτηση εκτός αιθούσης, ούτως ώστε να μπορέσει να λάβει το λόγο ο εισηγητής για το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψε για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Απασχόλησης όπου η κυρίως αρμόδια ηγετρία είναι η κυρία Όμιν Ρόιτεν. Είναι η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πράσινη Βίβλα για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά διεξοδικά συστήματα. This Έχει αναλάβει την έκθεση ο κύριος De Δεν βλέπω τους κύριους ηγητές, ο κύριος Έγκελ ήταν εδώ αλλά απεχώρησε. κύριος Κρότσμαν έχει πολλά ταλέντα και είναι εδώ. Δεν ξέρω τώρα από τους σοσιαλιστές ποιος είναι η κυρία Γκέπχαρτ. Εσείς είστε σκιώδης, μιλάτε αντί για τον σκιώδη. Όχι, λέει η κυρία Γκέπχαρτ. Και από βλάστον των πρασίνων, τέλος πάντων. Τότε θα κάνω εγώ τον σκιώδη συγκητή. Αλλά πρώτα πρέπει να ακούσω. Και θα πρέπει στις 5 να φύγω να πάω στην διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την Χρηματοοικονομική Κρίση. Πέστε με εγωμένως τη γνώμη της ε, Επιτροπής Ιστορικής Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι μια πρώτη ενέργεια απόψεων όπου θα πέσουν οι πρώτες προτάσεις και ιδέες. Και ε, er eh, μέχρι τις 16 του μηνός θα έχω προετοιμάσει τις τροπολογίες. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή τον Ιανουάριο και στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Συζήτησα με την κυρία Ούμαν Ρόιτερ και αν κατάλαβα καλά ε, ήθελε να επικεντρωθούμε στην ε, κατάσταση της εσωτερικής αγοράς δηλαδή την εσωτερική αγορά και ε, την ε, δυνατότητα επιλογής των εργαζομένων. Υπάρχουν και ε, πιο δύσκολα θέματα, η μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ε, και το ένα θέμα είναι η κρατική σύνταξη το οποίο έχει ρυθμιστεί παρόλο που υπάρχουν ακόμη ε, προβλήματα σχετικά με τις προθεσμίες της πενταετίας αλλά όταν πρόκειται για συντάξεις που βασίζονται σε συλλογικές συμβάσεις ε, το 2007 ήδη είχε διατυπωθεί μια νέα πρόταση και όλα αυτά ε, κόλλησαν από ό,τι κατάλαβα στο Συμβούλιο και ε, γι' αυτό υπάρχουν πολλά προβλήματα, το φορολογικό, διότι ε, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου, αλλά εάν καταβληθεί διασυνοριακά, σε ορισμένες χώρες υπάρχει φορολογική απώλεια ε, ε, υπερβολική ε, ε, παρακράτησης φόρων, οπότε όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα στο θέμα των συντάξεων και της αλληλεγγύης που θα πρέπει να τις διέπει και επ' αυτού θα πρέπει να εξετάσουμε τα διάφορα προβλήματα τα οποία τίθενται. Τίθενται προβλήματα και για την εσωτερική αγορά, δηλαδή και οι εργαζόμενοι έχουν προβλήματα εάν μετακινηθούν από το ένα κράτος στο άλλο και ίσως δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους τους τα, δικαιώμα, τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει πιο συγκεκριμένες προτάσεις και να μας πει συγκεκριμένα ποια προβλήματα υπάρχουν και τι προτείνει. Ε, το δεύτερο μέρος είναι πιο απλό. Ε, ε, δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι υπάρχει ένα σύστημα όπου δεν ξέρουμε ε, αν ε, παντού υπάρχει εξίσου καλή ρύθμιση και γι' αυτό είναι πολύ βασικό στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μην βασιστεί κανείς στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά να μειώσουμε την γραφειοκρατία και να μεγαλώσουμε τη διαφάνεια. Δεν, ε, δεν ε, προωθώ λοιπόν το θέμα της γραφειοκρατίας αλλά θα ήθελα να υπάρξει ελευθερία παροχής υπηρεσιών και βλέπουμε όταν συζητάμε με εργαζόμενους σε διασυνοριακές επιχειρήσεις ότι υπάρχουν προβλήματα. Ε, υπάρχουν και κοινωνικές διαφορές, ε, διαφορές στην κοινωνική ασφάλιση, στην ε, φορολογική νομοθεσία και δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιληθεί. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε και επιπλέον κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή πραγματεύεται και πιο γενικά θέματα. Χρειάστηκε να καταρτήσουμε μία γδομοδότηση και τέθηκε πάλι το θέμα εάν υπάρχει ένα υφόρο σύστημα συνταξιοδοτικό ή στα κράτη-μέλη διότι με τη γύρανση του πληθυσμού υπάρχει το πρόβλημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή τα κράτη τα οποία έχουν ένα σύστημα pay as you go θα αντιμετωπίσουν τα πιο σοβαρά προβλήματα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε ε, το σύστημα της εξοικονόμησης κεφαλαίων και ε, της αποταμίευσης και εκεί υπάρχουν λιγότερα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν και στο σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συντάξεις θα είναι αηφόρες πρέπει όμως να δούμε πόσο πρέπει να προχωρήσουμε διότι ε, χρειάζεται να υπάρξει αποταμίευση χρημάτων διότι ο πληθυσμός γυράσκει και μεταξύ των ε, παλαιών κρατών μελών υπάρχουν προβλήματα και ξέρουμε ότι οι συντάξεις ίσως δεν έχουν υπολογιστεί επακριβώς και στην ομάδα εργασίας του κυρίου ο Ρόμπο, θα ήθελα να ξέρω έχουν ληφθεί υπόψη τα θέματα αυτά ή όχι διότι αυτό που είναι βασικό ε, είναι να διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται όλο και περισσότερο ίσως αυτό μας απασχολήσει περισσότερο για τις γυναίκες και θα πρέπει ίσως η κατάσταση των γυναικών να είναι καλύτερα, καλύτερη και επιπλέον υπάρχει το θέμα των γνώσεων. Εάν δηλαδή οι γυναίκες είναι πιο μορφωμένες, πιο εκπαιδευμένες θα μπορούν να εργαστούν και περισσότερα και να προσχωρήσουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα πιο αργά. Τι γίνεται λοιπόν με το σημείο αυτό. Ε, ήδη οι ρυθμίσεις έχουν αλλάξει αλλάξει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, αναταραχές στη Γαλλία, στην Ελλάδα και υπάρχουν και άλλα θέματα. Σε περίπτωση που μειωθούν οι συντάξεις θα υπάρξουν προβλήματα στα κράτη-μέλη ε, σχετικά με το στόχο του 2020 για την καταπολέμηση της στόχιας. Ε, πιστεύω ότι και εκεί έχει γίνει ένα λάθος και θα πρέπει να υπάρχει και μία τρίτη εναλλακτική, δηλαδή οι ε, ιδιωτικές ασφαλίσεις, αλλά το θέμα είναι αν οι, άνθρωποι θα θα μπορούν να πληρώσουν διότι οι μελέτες απέδειξαν ότι ε, οι ατομικές ασφάλειες είναι οι πλέον δαπανηρές. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Όσον αφορά την αηφορία των συντάξεων θα ασχοληθούμε εμείς ή θα ασχοληθεί η Επιτροπή Απασχόλησης. Ένα άλλο θέμα. Τι πρέπει να γίνει σχετικά με την ε, ε, ρευστότητα ε, και τη φερεγγιότητα των συστημάτων των συνταξιοδοτικών, διότι τα συνταξιοδοτικά τα μία αντιμετωπίζουν προβλήματα, κάθε ένα έχει τη δικιά του δομή και μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί να κάνει διαφορετικές προτάσεις αναλόγως των καταστάσεων και θα επανέλθουμε όταν θα τις έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμη εικόνα που μας δώσατε και νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, σε αυτό το οποίο μπορούμε να προσθέσουμε εμείς ε, στη γνωμοδότησή μας, διότι σαφώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός ε, λέξεων που μπορείτε να έχετε. Μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι μία γνωμοδότηση είναι πολύ πιο αποτελεσματική αν στοχεύσουμε σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι πιο σημαντικά για μας. Ε, έχουμε και τους και Η κυρία Γκέπχαρτ θα μιλήσει εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ο κύριος Κρόιτσμαν θα μιλήσει. Κυρία Ρούλε, θα μιλήσετε κι εσείς εκ μέρους των Πρατσίνων. και θα μιλήσω κι εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου σύντομα. Να κάνουμε ένα γρήγορο γύρο λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίως συμφωνώ τόσο μαζί σας. Ακόμη και αν είχαμε διάθεση και μάλιστα μεγάλη διάθεση ε, να ε, πέσουμε μέσα στην, στο θέμα της φερεγγιότητας των ταμείων ε, δεν είναι εφικτό και θα πρέπει να περιοριστούμε σε ό,τι είναι εφικτό στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Θα ασχοληθώ με δύο θέματα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, οι συντάξεις δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Οπότε πρέπει να θυμόμαστε ότι Εάν αυτή η Επιτροπή και ακόμη περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προσφέρει προστιθέμενη αξία επί του θέματος, αυτό δεν θα επιτευχθεί με το να μπει στις λεπτομέρειες των μεγάλων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν ανά χώρα έτσι όπως διαμορφώνει την κατάσταση, αλλά θα πρέπει μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να έχει μία σταθερή στάση και να διαπιστώσει διαπιστώσει διάφορα θέματα ε, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων διότι σε όλη την Ήπειρό μας έχουμε ένα πρόβλημα χρηματοδότησης των, ε, ε, των συντάξεων στο σύνολό τους που είναι δύσκολες και που μας απειλεί όλους. Οπότε λοιπόν, είναι θέμα δημοσιονομικό και μέσω δημοσιονομικού προβλήματος απειλείται και η τήρηση των διατάξεων του Σύμφωνου Σταθερότητας και γενικότερα τη μεσονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα τμήμα μόνο του ευρύτερου προβλήματος. Το πώς δηλαδή τα δημοσιοοικονομικά θα διέπονται από κάποια διαχείριση που προσδοκούμε κάποια στιγμή να υλοποιηθεί, αλλά είμαστε ακόμα μακριά Επίσης, πέραν των ε, δημοσίων οικονομικών, θα πρέπει να δούμε και ένα πρόβλημα το οποίο είναι κυρίως ε, φιλοσοφικό. Ε, είναι, είναι θέμα ασφάλειας, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος. Ότι δηλαδή, εδώ και κάποια χρόνια, κάποιος αρχίζει να δουλεύει, γίνεται 80, 90, και δεν μπορεί πια να, να δουλέψει. Και όχι με την απόλυτη έννοια ε, του, Όμως μιλάμε για μια στατιστική που καλύπτει 20, 30 ή περισσότερα χρόνια για ε, τις χώρες που μας απασχολούν για πάρα πολλές χώρες Ευρώπης και ε, πέρασε επομένως εντός του αιώνα και επομένως τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει από το που ξεκίνησαν τα εξωτικά συστήματα και ακριβώς αυτό το οποίο σήμερα το θεωρούμε σαν ένα κεκτημένο δικαίωμα και ότι κανεί θα πρέπει να απολάβει αυτού του δικαιώματος μόλις το θελήσει. Και πρόκειται αυτή τη στιγμή, όπω ξέρετε, για την προβληματική που απαιτείται στη Γαλλία, πρώτα για ένα βάρο που έχει μετακυληθεί στου πιο νέου στην κοινωνία. Και όλο ένα και περισσότερο απασχολεί τους Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες και δεν πρόκειται μόνο για την ενεργή περίοδο της σταδιοδρομίας, είναι το ότι όλο και περισσότερο η κατάρτιση παίρνει χρόνο, μετά μεγαλώνει η περίοδος ε, που κανείς είναι στη σύνταξη, επομένως και το Κοινοβούλιο αλλά και η Επιτροπή θα πρέπει να τοποθετηθούμε και να προσαρμόσουμε την προβληματική μας ανάλογα με τις μεταβλητές που υπάρχουν και να προχωρήσουμε αναλόγως στην θέση της κατάλληλης νομοθεσίας. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο η κυρία Ευχαριστώ. Και εγώ ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το σκιώδη συγητή που δεν ε, μπορεί να, ε, να παρασταθεί διότι είναι στο Παρίσι για μια σημαντική συνεδρίαση αλλά θα προσπαθήσω να τον εκπροσωπήσω. Ο κύριος De Jong έχει κάνει ορισμένα ερωτήματα, δηλαδή τι θα πρέπει να συζητήσουμε σαν Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών και αυτό είναι το πιο βασικό θέμα διότι όλα τα θέματα που αναφέρονται στις συντάξεις έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών δηλαδή ε, την προστασία των ανθρώπων όταν γερνάνε. Είναι δύσκολο λοιπόν να αποκλείσουμε κάτι που δεν θα ήταν στις αρμοδιότητές μας διότι όλα αυτά είναι σχετικά και αφενός πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι συντάξεις στα κράτη-μέλη και αυτό είναι θέμα ε, των κρατών μελών. Δεν μπορούμε εμείς ε, να επιληφθούμε, δεν έχουμε αρμοδιότητα, ε, είναι θέμα των κρατών μελών. Αλλά υπάρχουν όλο και περισσότεροι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ερώτημα είναι ποιες είναι οι απαιτήσει των συντάξεων, των επαγγελματικών συντάξεων, ε, πώς εξελίξονται οι συντάξεις αυτές εις ε, τον κόσμο που ζούμε και πόσο μπορούν να διαφυλάξουν οι ενδιαφερόμενοι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Και εδώ είναι το θέμα και το συντάξεων χειρίας ή εν πάση περιπτώσει ατόμων που έχασαν τα δικαιώματά τους διότι παντρεύτηκαν εκτός του κράτους τους και δεν έχουν πλέον δικαίωμα όχι για μας τους Γερμανούς, αλλά σε άλλες χώρες όπως διαπίστωσα. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στο θέμα αυτό. Δηλαδή να δούμε πώς όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Όταν λοιπόν κοιτάζω το, την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω ότι αυτά τα θέματα δεν συζητούνται σωστά διότι στην πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εξετάζουμε μόνο ένα ιδεολογικό θέμα σύμφωνα με το ρητό ότι έχουμε δημογραφικές αλλαγές και αυτές οι δημογραφικές αλλαγές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή οι άνθρωποι θα πρέπει να, ζουν να εργάζονται πιο πολύ καιρό για να μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Είναι μια πολύ κοντόφθαλμη απάντηση την οποία ε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διότι ε, δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις. Ε, πότε εγκαταλείπουν τον ε, χώρο της εργασίας ε, οι άνθρωποι βλέπουμε ότι είναι πριν από τα 60. Αν λοιπόν φτάσουμε στα 67 ή στα 70 που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το σύστημα των συντάξεων δεν είναι υλοποιήσιμο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να αλλάξει η χρηματοδότηση που θα πρέπει πρέπει να συμπληρωθεί με φορολογικούς πόρους. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς είναι δυνατόν ε, να επηρεάσουμε τη συζήτηση για τον ε, κόσμο που αλλάζει και στον οποίο ζούμε και να μην κοιτάμε μόνο το σημείο όπου ξεκινάει η σύνταξη γιατί είναι πολύ κοντόφθαλμο και δεν μπορούμε να απαιτήσουμε ε, οι άνθρωποι να εργάζονται μέχρι τα 80 τους τους. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ας δούμε πού μπορούμε να διατυπώσουμε απαντήσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα και να μην είναι απλώς θεωρητικές απαντήσεις που προσπαθούμε να δώσουμε. Από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Τώρα λίγο ξέφυγα από το θέμα μου, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς είναι δυνατόν στον επαγγελματικό κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα να διαμορφώσουμε τη σωστή χρηματοδότηση σε στα κράτη-μέλη. Γνωρίζω περισσότερο την κατάσταση στη Γερμανία από τις άλλες χώρες. Εάν λοιπόν παρακολουθήσω τα ταμεία των ελευθέρων επαγγελμάτων όπου δεν υπάρχουν και δεν δημιουργούνται αποθέματα όταν βλέπω ότι το κράτος για τους δημοσίους υπαλλήλου δεν δημιουργεί αποθέματα, αποθεματικά, τότε ίσως στο θέμα της χρηματοδότησης υπάρχουν σημεία τα οποία πρέπει να εξετάσουμε προτού εξετάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται επαγγελματικά και δούμε πώς μπορούμε να βρούμε άλλες λύσεις. Και σαν Ευρωπαίοι πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορούν να δοθούν ενάυσματα στα κράτη-μέλη για να αλλάξουν οι όροι συνταξιοδοτήσεως κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι αλλαγές να μην γίνουν εις βάρος των εργαζομένων πράγμα το οποίο εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς αλλά πώς μπορεί ολόκληρη η κοινωνία να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των συντάξεων ώστε να γίνει αυτή εφικτή. Ε, βλέπω παραδείγματο χάρη ότι ο κύριος Έγγελ είχε πει στην αρχή ότι πρέπει να περιορίσουμε και μετά άνοιξε ε, πολύ το θέμα και εγώ άφησα μία πτυχή των σκέψεών του γιατί νομίζω θα πλατιάζαμε πάρα πολύ αλλά πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε σφαιρικά και να μην εξετάσουμε ε, στιγμιαία ορισμένα σημεία και ε, βλέπω ότι ε, δεν συμμετέχει η Επιτροπή Ελευθεριών που θα μπορούσε να καλύψει τη σκοπιά των δικαιωμάτων του πολίτη. Ε, σαν όμως Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προσπασίας των Καταναλωτών είμαστε αρμόδιοι και θα πρέπει ίσως να ενισχύσουμε τη σκοπιά της προστασίας των καταναλωτών και να φροντίσουμε ώστε οι άνθρωποι όταν γεράσουν να μπορούν μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και το δημόσιο να μπορέσει να εξυπηρετήσει αξιοπρεπώς τους πολίτες. Είναι βέβαια τετραγωνισμός του κύκλου, αλλά πρέπει όλα να τα πετύχουμε. Τι να σας πω. Θα πρέπει να μου επιτρέπετε κύριε γιατί θα πρέπει να πάω. Ε, γίνεται συνδυασία για την κρίση, γιατί ε, αφορά το κομμάτι της δικής μας ομάδας και τώρα ο κύριος Τριανταφυλλίδης θα με ε, διαδεχθεί στην Προεδρία, φαντάζομαι ότι πάρα πολύ καλά θα προεδρεύσει. Κυριάκο, αν θέλεις, έλα να προεδρεύσεις για μένα, αλλά, αλλά πρώτα, επειδή είμαι ο σκιωδησηγητής της ομάδας, έλα, οπότε δεν θα υπάρχει διακοπή στη διαδοχή. Στον πρώτο όροφο, στο πρώτο επομένως ε, στο, στην αίθουσα υπαριθμών 1 γίνεται αυτή η συνεδρίαση και ε, θα είναι τη Διακυβευτική ε, Επιτροπή για την κρίση και θα συνεδρίσω του Ούγγρου συναδέλφου. Δεν πρέπει να αργήσω. Όμω, έχω τα εξή να σα πω από πλευρά μου έχει δίκιο η κυρία Γκέμπχαρτ. Όλα αυτά αφορούν και την ιστορική αγορά. Να δούμε εμείς πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην προβληματική. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών πρόσφατων και αυτό εξαρτάται από το πόσο θέλει και μπορεί κανείς να ασκήσει το επάγγελμά του σε διαφορετικές χώρες. Εάν διαπιστωθεί ότι τα, στα εξωτερικά τους δικαιώματα αποτελούν πρόβλημα για το σκοπό τους αυτό, γιατί πρέπει να καταλήξουν το εθνικό του σύστημα στη εξοδότηση και δεν μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματα, τότε έχει κάνει ένα συμφέρον να κάνει κάτι ώστε να λειτουργήσει όπως πρέπει η εσωτερική αγορά και άρα αυτό είναι πρόβλημα. Είναι μια πρόκληση για την εσωτερική αγορά. Είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πολιτικής για την καινοτομία και οι ερευνητές. Επομένως, Θέλουμε να μπορούν να πάνε από τη μία χώρα στην άλλη, θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο να βοηθούν. Έχει προσπαθήσει μόνο σε διάφορε χώρε και να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω κινητικότητα δεν υπάρχει ενώ θα έπρεπε. Κάτι εξοχή να υπάρχει για αυτού του ανθρώπου. Να το προσέξουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξή. Το συνταξιδοτικό είναι περίπλοκο πρόβλημα για τους καταναλωτές. Κυρίως λόγω της σχετικής νομοθεσίας και τα ξέρετε. Τα ξέρετε και επομένω. αυτό που σημαίνει κανείς να έχει τη γνώμη του ειδικού. Σε πολλές περιπτώσεις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα έχουν συνέπειες όταν κανείς παίρνει σύνταξη του από 20-30 χρόνια. Αυτό αφορά και την καταναλωτική πίστη, είπαμε. Θα πρέπει κανεί να μπορεί να έχει συμβουλού ανεξάρτητους και αμερόληπτους και το έγγραφο της Επιτροπής αναφέρεται το ότι θα πρέπει να υπάρχει και στις σε ενιαία αγορά. Και εδώ υπάρχουν θέματα αυτό είναι αρμόδια δική μας, όχι αρμόδια της Οικονομικής Επιτροπής και τους είπαμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε πάρα πολύ σωστά τα λέει ο κ. Ντεγιόν. Για το time share και για άλλα θέματα τα οποία έχουμε μελετήσει. Νομίζω ότι έχει υπάρξει προσθέμενη αξία. Και όσον αφορά τα στοιχειωτικά ταμεία, τη ρευστότητα αυτών. Βεβαίω υπάρχουν κυρίως αρμόδιες επιτροπές που είναι άλλες από τη δική μας, αλλά έχουμε και θέματα εδώ που μας αφορούν. Και άρα μπορούμε επί του προκειμένου να βοηθήσουμε την Επιτροπή Απασχόλησης. Όλα αυτά επομένω θα πρέπει να υπόψη από τον κύριο Ντεγιόν και τώρα τη σκητάλη στον Κυριάκο για να προεδρεύσει για την υπόλοιπη συνεδρίαση. speaker Mr. You have the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το, η πράσινη βίβλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αναφέρεται στα ευρωπαϊκά συστήματα και πιστεύω ότι σε πολλά ε, σημεία είναι σωστή. Πρέπει να δούμε όμως τι, πώς θα προχωρήσουμε, διότι αφενός Υπάρχουν τα συστήματα τα συνταξιοδοτικά στα διάφορα κράτη, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα χρηματοδότησης. Στην ε, Γερμανία πληρώνουν οι εργοδότες, οι ε, εργαζόμενοι, αλλά ε, συμβάλλουν και οι φόροι σε ορισμένα κράτη. <coughs> Οπότε το ερώτημα είναι αν θέλουν ορισμένοι να αλλάξουν τα συστήματα αυτά όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορούμε να επέμβουμε. Υπάρχουν διάφορες προσφορές και ε, μπορούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Ο κύριος Ντεγιόγκ όμως μας είχε πει, τι, μας είχε ρωτήσει επίσης τι θα γίνει και με τις ε, επιχειρησιακές συντάξεις. Υπάρχουν και ε, οι θέσεις των ε, εργαζομένων. Οπότε, αν πρόκειται για συνταξιοδότηση από μία επιχείρηση, θα πρέπει να δούμε τι προβλέπει η οργάνωση του συστήματος και υπάρχουν διάφορες μορφές αναλόγως της νομοθεσίας και αναλόγως της χώρας και γι' αυτό οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να ισχύσουν διασυνοριακά και αυτό είναι πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να προβούμε σε αλλαγές διότι ε, στην ε, Ευρώπη υπάρχει ε, μία ενιαία αντιμετώπιση ως επιτοπλίστων και δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Αυτό που είναι πιο επικίνδυνο είναι οι διαφορές ισορροπιών σε διάφορα κράτη μεταξύ συντάξεων του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και προοπτικών διότι μία ε, ενίσχυση των απαιτήσεων ιδίου κεφαλαίου θα οδηγούσε ε, σε ε, επιμήκυνση του χρόνου εργασίας και θα διακινδύνευε το σύστημα διότι αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών ε, συστημάτων ενδέχεται ε, να σταματήσουν να συμβάλλουν διότι ε, δεν θα θέλουν να χρηματοδοτήσουν άλλους και να πληρώσουν περισσότερα. Οπότε πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην διακοπούν οι εισφορές. Και όπως σας είπα μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν μεγάλες διαφορές και όταν κοιτάμε τα συστήματα που αναφέρονται στις συντάξεις των επιχειρήσεων υπάρχει θέμα σχετικά με τη χρηματοδότηση. Ε, τώρα έχουμε πρόβλημα με την γύρανση του πληθυσμού και αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν σήμερα μειώνονται όλο και περισσότερο σε ορισμένα κράτη-μέλη και η αναμονή ζωής ε, των ατόμων αυξάνεται όλο και περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν μια ανισορροπία την οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε και πρέπει να δούμε αν θα επιτευχθεί ή όχι είναι, ε, ε, είναι όμως ένα σημείο που μας απασχολεί. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στη Γερμανία και πόσο προσπαθεί κανείς να χρηματοδοτήσει αυτές τις ανισότητες και γι' αυτό θα πρέπει ε, να μην διακινδυνεύσει ο τρίτος πυλώνας που είναι η συντάξη των επιχειρήσεων και να μην μας απασχολήσει να το αποκλείσουμε δηλαδή το θέμα αυτό από τη συζήτηση τώρα. Thank you, Mr. Kreutzmann. And uh, the floor goes to Mrs. Rule. Μία σύντομη ηρωνική παρατήρηση. Εις, ε, τις ε, εφημερίδες ε, σχετικά με τη συζήτηση ε, για τις ε, συντάξεις ε, λέχθη στις εφημερίδες ότι εφόσον είναι τόσο πλουσιοπάροχη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συντάξεις του δικού της προσωπικού και των επιτρόπων δεν είναι σε θέση να μας δώσει συμβουλές σε εμά τους εκτός. Ουσιαστικό όμως, όπως είπε και η κυρία Γκέπχαρτ, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν δύο θέματα που πρέπει δύο να μας απασχολήσουν. Καταρχήν το θέμα της κινητικότητος και δεύτερον το θέμα της διαφάνειας. Δηλαδή θα πρέπει όλοι οι πολίτες να τύχουν μιας καλής υπηρεσίας θα ζητήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και δεν νομίζω ότι στο σημείο αυτό προσκρούμε στην επικουρικότητα, αντιθέτως. Και η άλλη παρατήρηση που κάνατε ε, κύριε Κρόιτσμαν δεν είναι αρμοδιότητος της δικιάς μας Επιτροπής αλλά της Οικονομικής Επιτροπής. Εμεί θα πρέπει ιδίω ε, να δούμε ε, αν μπορεί κανείς ε, να μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα και αν μπορεί να αυξήσει την διαφάνεια. Υπάρχει ακόμη κάποιο που έχει εγγραφεί να λάβει το λόγο, που είναι ο κύριος Ζουβάν και κατόπιν θα λάβει το λόγο ο κύριο Ντεγιόν. Ζουβάν, ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλά ήδη αναφέρθησαν, αλλά θα πρέπει πρώτα πρώτα να τονίσουμε αυτό το οποίο είπαν πολλοί ότι δηλαδή η πολιτική τη σύνταξη είναι κάτι το οποίο προσυδειάζει στο κράτο. Οπότε, αφού ασχολούμαστε με αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Τέσσερα σημαντικά σημεία, να σα αναφέρω ταχύως. Πρώτα απ' το, το σύστημα θα πρέπει να διακρίνεται από ε, ε, διαφάνεια και να είναι και κατανοητό. Το είπαν πολλοί συνομιλητέ. θα πρέπει κανεί να καταλαβαίνει τα δικαιώματά του για να μπορέσει να τα ασκήσει. Και ακριβώ το δικαίωμα στη σύνταξη επίση πρέπει να είναι κατανοητό. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να λέμε ψέματα ούτε διαπαραλήψεις, διότι σήμερα τα συντηρησιωτικά συστήματα όπως και είναι οργανωμένα περνάνε από πάρα πολύ δύσκολες ώρες από πλευρά οικονομικής και δεν είναι και πάρα πολλά για τα σενάρια ή θα πρέπει κανείς να ε, δουλεύει πιο μεγάλο χρονικό διάστημα για να έχει περισσότερες ε, εισφορές ή θα πρέπει κανείς να αυξήσει τις ε, εισφορές ακριβώς όπως αναφέρθηκε. Όμως, όπως είπε η κυρία Γκέπχαρτ, δεν θα πρέπει να κολλάμε μόνο στο θέμα του ηλικιακού ορίου. Είναι σημαντικό, έχετε δίκιο. Όμως το να λέμε ότι η ηλικία είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημασία και αυτό δεν είναι ειλικρινές. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις τρεις αυτές μεταβλητές. Θα πρέπει επομένως οι πολιτικοί να αποφασίσουμε ε, ποια, μεταβλητή θα ρίξουμε το, το ειδικό μας βάρος. Απ' την άλλη μεριά, κάθε μεταρρύθμιση θα πρέπει να διακρίνεται από δικαιοσύνη σχέση μεταξύ των γενναιών. Δεν θα πρέπει να επιβαίνουμε κάποιου οι οποίοι ε, αύριο θα πάρουν λιγότερα από όσα έχουν εισφέρει. Επίση, θα πρέπει όλοι να απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων ε, ανάλογα με το πόσο έχουν δουλέψει. Επίσης, εάν το σύστημα δεν προσαρμοστεί, πρόκειται να φτωχεύσει. Και επίσης, το ίδιο αφορά και τις επικουρικές συντάξεις. Πολύ σημαντικό. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι εάν το βασικό θέμα δεν επιληθεί με αλληλεγγύη, τότε κάποιοι θα μπορέσουν να έχουν σύνταξη, αυτοί μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές για την επικουρική σύνταξη. Είναι μια για το οποίο το κληροδοτούμε η μια γενιά στην άλλη το συνταξιωτικό δικαίωμα και να προσέξουμε αν υπάρχει μια, μια ανισότητα, δηλαδή ότι αυτοί που έχουν τα λιγότερα χρήματα, αυτοί που θα έπρεπε να καλυφθούν, αυτοί να δικαιωθούν και μην έχουν σύνταξη. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή του συστήματος. Κύριε Ντεγιόγκ, εσείς για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, διότι θεωρώ ότι έδειξε αυτή η συζήτηση το τι θα προκύψει για την Επιτροπή της Απασχόλησης. Τα είπα και στην εισήγησή μου ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα θέματα εσωτερικής αγοράς. Μάλκομ Χάρμπορ ανέφερε κάποια θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Η συζήτηση, το θέμα είναι τεράστιο. Το ηλικιακό όριο, τα δικαιώματα εν γέννη, τα στεξιωτικά. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημαίνει η δική μας αρμοδιότητα. Θα πρέπει θα αρχής να το ξεκαθαρίσουμε γιατί ακούμε ένα σωρό επιχειρήματα και εγώ έχω απόψη για όλα αυτά δεν είπα τίποτα. Γιατί όλα αυτά θα ζητηθούν θα είναι στο επίκεντρο συζήτηση στην Επιτροπή Επασχόλησης. Αλλά ασχοληθούμε με το θέμα της αγοράς. Τη διαφάνεια, να, πώς είναι κατανοητό το σύστημα και να κάνουμε και κάποιες γενικές διαπιστώσεις. Η γνωμοδότηση αυτή θα είναι σύντομη, αλλά έχουμε και το θέμα αυτού που προανέφερα του τρίτου πυλώνα και να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει ποιοι είναι οι φραγμοί στα προγράμματα στις ιδέες που αφορούν τον τρίτο πυλώνα. Όλα αυτά θέλω να τα συνοηθώ, να τα ξεκαθαρίσω με τους κοιόδες ηγητές και έτσι να βγει μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας από όλα αυτά. Thank you, Mr. De Jong, and thank you to... Ευχαριστούμε κύριε Δεγιόγκ και ευχαριστώ και σε όλους τους ομιλητές. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι τα διάφορα. Έχει κάποιος κάτι από τα διάφορα. Αν όχι, Επόμενη συνεδρίαση αύριο στις 3. Ε, Φόρουμ για την ενή αγορά. Ευχαριστώ.